από όλους κοινό, από κοινό. Για τα πρακτικά της 27 Μαΐου 2015 έχετε στη διάθεσή σας τα πρακτικά. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Ο κύριος Γκλέζος θέλει το λόγο για τη μερίσια διάταξη. Αγαπητέ Πρόεδρε, λυπούμε ιδιαίτερα που είμαι υποχρεωμένος και πάλι να αναφερθώ σε εσά προσωπικά. Πριν από λίγο ακούσαμε έναν ωραίο ρητορικό λόγο που ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα σχετικά με τα διδατορικά καθεστώτα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Όμως σήμερα η ελεύθερη Ελλάδα μια χώρα που εκφράζει τη βούληση του ελληνικού λαού για να χαράξει τη δική της πορεία συναντάει την σφοδρή αντίδραση από την πλευρά των τριών θεσμών τρόικα και από την πλευρά τη δική σας και μου κάνει εντύπωση με ποιο δικαίωμα ως πρόσωπο έχετε δικαίωμα να επέμβετε να πείτε οτιδήποτε αλλά ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νομίζω ότι δεν έχετε το δικαίωμα να εκφράζετε το, το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να επεμβαίνετε στην Ελλάδα και να προσπαθείτε να την στραγγαλίσετε. Μακριά τα χέρια όλων των δανειστών από την Ελλάδα. Θα είναι γελασμένοι όσοι νομίζουν ότι θα υποτάξουν τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ντούντα